Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την κοινή συνάντηση ΦΕΜ e και ΙΝΤΑ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ και της Επιτροπής ΦΕΜ e σε αυτήν την κοινή συνάντηση. Είναι χαρά μου που συμπροεδρεύω με τον Γιούλιο Βίγκλερ, τον αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής. Ήταν ένα σημαντικό φάκελο για τις δύο επιτροπές. Θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων ως ε, μια βασική αξία της Ένωσης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στην εμπορική πολιτική. Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε λοιπόν από αυτή του φακέλου κατά τη διάρκεια της κοινή ακρόασης που έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια είχαμε τη δυνατότητα ε, να διαπιστώσουμε ότι οι συμφωνίες, οι εμπορικές και οι επενδυτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για τις άντρες και τις γυναίκες. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να αναλύσουμε τη νέα εμπορική πολιτική από μια προοπτική ισότητα των δύο φύλων. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίγκλετ ω εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, να καλημερίσω και τα μέλη της Επιτροπής ΦΑΜ και της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι τιμή μου που εκπροσωπώ την Επιτροπή μου την ΙΝΤΑ σε αυτή τη κοινή συνεδρία σήμερα για να συνεχίσουμε να συζητάμε για την ισότητα των δύο φύλων στις εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή, Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2015 έδωσε έμφαση σε μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται στι ευρωπαϊκέ αξίε. Φτάνουμε στην πρώτη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νέα εμπορική στρατηγική τη, τον Νοέμβριο φέτο. Η ε, Επιτροπή, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα οργανώσει μια συνάντηση όπου θα συζητηθεί αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ υποστηρίζει βεβαίω μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται στι αξίε μα και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ ζητούμε και εμεί όταν των δύο φίλων στι εμπορικέ μα συμφωνίε ως μια αρχή, ως ε, ε, ένα στοιχείο που πρέπει να διέπει τι πολιτικές μα. Έχουμε ζητήσει μια ε, πραγματονομοσύνη, δύο μελέτες μάλλον, ε, για την εμπορική πολιτική από την εθελοτυφλία συστήματα ισότητας των δύο φύλων σε μια ευαισθησία ε, έχουμε ζητήσει και μια άλλη μελέτη από εξωτερικούς συνεργάτες. Φτάνουμε τώρα στα συμπεράσματα. Θέλουμε να βοηθήσω, θέλω να ευχαριστήσω μάλλον το, τον εισηγητή, τους εισηγητές και τους χειόδες εισηγητές για το έργο τους και ελπίζω η σημερινή συζήτηση να συνεισφέρει για να οδηγηθούμε σε μια ισορροπημένη, ρεαλιστική αλλά και καινοτόμο προσέγγιση στα πλαίσια της ε, ε εκθέσεις αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εισηγητές η κυρία Μπιόρκ. Τώρα θα μιλήσετε εκ μέρους και των δύο εισηγητών, να κατάλαβα καλά. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της συναδέλφου, αλλά είχε ένα πρόβλημα τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να φύγει από την Ιταλία σήμερα το πρωί. Η κυρία Φορέντσα. Θα μιλήσω στα σουηδικά, οπότε όποιος χρειαστεί παρακαλώ να φορέσει τα ακουστικά του, λέει ο μιλητρία. Συνεχίζω λοιπόν. Η γνωμοδότηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εγώ θα ήθελα από την αρχή να εξηγήσω ότι η Επιτροπή Γυναικών θεώρησε σημαντικό να ασχοληθεί με μια γνωμοδότηση της ισότητας των φύλων στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών. Και με χαρά μάθαμε ότι και η Επιτροπή ήθελε να συμμετάσχει ε, στη δουλειά αυτή, στην προσπάθεια αυτή. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ Σήμερα ήμουνα σε επαφή και με τα μέλη της ΔΕΒΕ για να υποβάλω το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης. Είχα και τα πρώτα σχόλια και παρατηρήσεις από πλευρά τους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνεργασία ΚΙΜ μαζί τους. Είναι μια σημαντική προοπτική αυτή επίπεδο μάλλον ε, εκείνο της ισότητας των φύλων στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών Έχουμε πλέον διοργανώσει ακροάσεις ε, ε, για να ακούσουμε και ενδιαφερομένους φορείς ε, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με εμπορικούς εταίρους. Πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρόκειται για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν τεράστια σημασία και αντίκτυπο. Επομένως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, υπόψη και οι στόχοι μας στα κοινωνικά πλαίσια και πλαίσια ισότητος των φύλων και ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει επαναλάβει επανειλημμένως ότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, και συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών έχουμε πάρα πολλές και διαπραγματευόμαστε πάρα πολλές ακόμα. Όλες αυτές θα πρέπει να τις διαπραγματευόμαστε επί τη βάση και των αρχών μας που συμπεριλαμβάνουν την ισότητα των φύλων. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης αυτής, της γνωμοδότησης αυτής, περιμένουμε τα σχόλιά σας εμείς ε, διαιρέσαμε το σχέδιο σε ε, κάποια κεφάλαια, ένα που είναι πιο γενικό αν θέλετε, ευρύτερο, δηλαδή οι προοπτικές ε, των θέματων ισότητας των φύλων στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες, ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά συγκεκριμένους τομείς εμπορικούς και οικονομικούς και είμαι σίγουρη ότι και με τη δική σας βοήθεια, με τις δικές σας παρατηρήσεις και σχόλια και μαζί με τα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε και κεφάλαια ή παιδεία που ακόμα ενδεχομένως να μην έχουμε συμπεριλάβει. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι οι γνωμοδοτήσεις ε, που θα υποβάλουμε στο μέλλον ε, σε σχέση με ακριβώς με διεθνείς συμφωνίες. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα στοιχεία της νομοδότησης. Δεν πρόκειται να αναφέρω το σύνολο, αλλά ε, σημειώσαμε και υπογραμμίσαμε ότι λείπει το πεδίο, η προοπτική της ε, υποστήριξης της ισότητας των φίλων. Μιλούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να έχουμε μια στρατηγική με συγκεκριμένα μέσα υλοποίησης. Και αυτό σχετίζεται με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τους εκπροσώπους ε, της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας σε εμπορικό επίπεδο αναφερόμενοι στις διάφορες συμβάσεις που έχουμε επικυρώσει όπως εκείνη για την ε, ε, εκρίζωση όλων των διακρίσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην αγορά και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εισαχθούν στο πλαίσιο της εμπορικής μας πολιτικής. Λέμε στην κοινομοδότηση ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη γνώση για τα θέματα ίσων ευκαιριών όταν διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες υπό την οπτική των γυναικών γιατί πολύ συχνά βλέπουμε αρνητικές συνέπειες, αντίκτυπο που προκύπτει, που απορρέει από την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση δημοσίων φορέων. Πώς λοιπόν επιδρά αυτό, τι αντίκτυπο έχει επί του γενικού πληθυσμού. ναι ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι ένα χρήσιμο μέσο οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που εμείς όλοι εδώ προσυπογράφουμε και υπερασπιζόμαστε. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα δεσμευτικά πρότυπα στα πλαίσια της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. γιατί είδαμε και πόσο δύσκολη ήταν η συζήτηση σχετικά με, την, με το διεθνής δίκαιο και τον σεβασμό συγκεκριμένων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες ζώνες. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ώστε όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισμοί μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, μαζί με τον ΠΟΕ να έχουμε κοινέ στοχεύσεις και κοινέ προθέσεις θα μείνω εδώ, αλλά περιμένω, περιμένουμε τις χρήσιμες παρατηρήσεις σας, ώστε αυτή η γνωμοδότηση να εμπλουτιστεί και να είναι όσο γίνεται πληρέστερη. Είναι σημαντικό να εργαστούμε προκειμένου να δείξουμε στην Επιτροπή ότι είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυτό που επιδιώκουμε. Να έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο επίπεδο επίγνωσης ε, των θεμάτων ισότητας των φύλων στα πλαίσια των διεθνών εμπορικών μας συμφωνιών. Περιμένουμε τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση και τώρα θα στραφώ στους κοιόδης εισηγητές από την Επιτροπή ΦΑΜ. Ε, δεν πρόκειται να σεβαστώ τη σειρά διότι ο κύριος Ρόντορ που πρέπει να φύγει ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Βεβαίω, στι 5 πρέπει να πάω στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο πρώτο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο εισηγήτριες ε, για την εργασία τους για αυτό το επίκαιρο θέμα. Όπως ξέρουμε θα πρέπει κατεπηγόντως να ε, ασχαληθούμε ε, με την τυφλότητα σχετικά με τα φύλλα της εμπορικής πολιτικής έχουμε το εμπόριο για όλους, η στραγική αυτή δεν αναφέρει καν την ισότητα των φύλων με αυτές τις εκθέσεις. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι το εμπόριο δεν είναι ουδέτερο ως προς το φύλο και να δούμε πώς θα μετρήσουμε τον αντίκτυπο και θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία ασχολείται με τον σύγχρονο ρόλο των φύλων θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές ιδέες που μπορεί να είναι χρήσιμες για την εργασία μας. Πρέπει να αναφερθούμε ε, στις εντολές των, ε, τις διαπραγματευτικές στην έλλειψη των θεμάτων σχετικά ε, με τα φύλλα. Τα φύλλα ερμηνεύονται με τρόπο στενό ή λείπουν από την, τον αντίκτυπο, την μελέτη αντικτύπων και οι μελέτες αυτές, οι αξιολογήσεις θα πρέπει να δούνε τη δυναμική που υπάρχει σε σχέση με τις αλλαγές και να έχουν μια προσέγγιση συστημική και συνολική. Πριν από κάθε συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση του αντικτύπου. Έχουμε επίσης να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει ε, για όλες τις ε, διαφορές ε, να υπάρχει ένα κεφόλαιο σχετικά με την ισότητα των φύλων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν δεδομένα για να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν πάνω στις γυναίκες οι συμφωνίες και στην ισότητα των φύλων και να ορίσουμε ένα κομβικό σημείο μέσα στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για να υπάρχει ένα mainstreaming στην εμπορική πολιτική. Η Κομισιόν θα πρέπει να, ε, να εκπαιδεύει τους διαπραγματευτές και τους αξιωματούχους. Πρέπει επίσης οι να αναφερθούμε σαφώς στο γεγονός ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και αυτό ε, μπορεί να υπονομεύσει την δίκαιη παροχή των υπηρεσιών διότι οι γυναίκες είναι οι βασικοί φροντιστές ε, της κοινωνίας μας. Νομίζω θα πρέπει να ζητήσουμε ε, την μετάλλαξη, την μεταμόρφωση όλων των πολιτικών και εργαλειών για να προωθήσουν την ισότητα και την δικαιοσύνη μεταξύ των φίλων. Αυτές είναι οι ιδέες που θα χαιρόμουν να συζητήσω με τις εισηγήτριες. Έχω την πλήρη υποστήριξη των όσων, ε, έχουν την πλήρη υποστήριξη των όσων παρουσίασαν και θα έχουμε νομίζω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για το μέλλον. Ευχαριστώ για την κατανόηση και τώρα η κανονική σειρά ΦΕΜ σκιωδών εισηγητών για το ΕΛΚΑ ε, τα σημεία της Μπάρμπαρα Μαντέρα θα παρουσιαστούν από τον Σαλβατόρη Τσίκου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, η κυρία Ματέρα Σκιώδης ε, του ΕΛΚΑ ε, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω ε, και ζητάει συγγνώμη που δεν μπορούσε να είναι εδώ παρούσα σήμερα. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τις εισηγήτριες, τις κυρίες Μιγιόρ και Φορέντσα. Είμαστε πεπισμένοι ότι το πεδίο του διεθνούς εμπορίου και αυτές οι πολυμερείς διεθνείς εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες μπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την ε, ενίσχυση της οικονομικής θέσης των γυναικών. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράγματι, θεωρούμε, κάποιες πτυχές των συμφωνιών αυτών για να βελτιώσουμε την κατάσταση στις χώρες εκείνες όπου έχουμε ακόμα σημαντικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην Επιτροπή Γυναικών έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ανεπαρκή συνένεση επί των μεθοδολογιών λεπτομεριών ενσωμάτωσης των στοιχείων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να μπορούν ισότιμα να επωφελούνται των θετικών στοιχείων των συμφωνιών αυτών των εμπορικών δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να αναλύει κανείς από τις πρώτες φάσεις, από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, ε, τον αντίκτυπο επί των ανδρών και γυναικών ανεξαρτήτως ιδεολογικής προσέγγισης. Και αυτά ισχύουν για όλες τις περιφέρειες του κόσμου, για όλες τις χώρες του κόσμου, αυτά τα προβλήματα δηλαδή, το οποίο είναι απαράδεκτο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης αξία και ιδρυτική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίζουμε αυτό στα πλαίσια της ε, υπογραφής οποιασδήποτε εμπορική συμφωνίας. Κάποιες από τις δηλώσεις που γίνονται και κάποιες από τις πιέσεις που ασκούνται ενδεχομένως είναι υπερβολικά ιδεολογικά φορτισμένες. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο σχέδιο, στην γνωμοδότηση, να δώσουμε ένα πιο ισορροπημένο χαρακτήρα φαίνεται να ηχνηλατείται να διαγράφεται στο κείμενο μια τάση εξωστρακισμού κάποιων φαινομένων, χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκείς παραθέσεις και αναφορές. Έχουμε ομάδες πληθυσμού που επωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο, αλλά το να λέμε γενικώ και ορίστως ότι όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες, χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, δεν μας βρέχει σύμφωνος. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει στις εμπορικές συμφωνίες να δοθεί μία επιπλέον διάσταση συμμετοχικότητος και ισότιμης μεταχείρισης και ευκαιριών χωρίς διακρίσεις χωρίς διακρίσεις μεταξύ πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών των τρίτων των πολιτών, με συγχωρείτε, των τρίτων χώρων με τις οποίες διαπραγματευόμαστε, γιατί εξάλλου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται την ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλα τα πεδία της αγοράς, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνο να έχει το ρόλο του επιμορφωτή πρέπει να καταβάλει και μια ελάχιστη προσπάθεια προς την κατεύθυνση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κάθε κατάκτηση πρέπει να αξιολογείται σωστά και κάθε δυνατότητα επίτευξης θετικού αποτελέσματος πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιό της. Όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν αυτόματα άμεσα σε ένα βήμα ώστε άλλες τρίτες χώρες να φτάσουν στα δικά μας υψηλά επίπεδα κοινωνικών κατακτήσεων. Δηλαδή το να σκεφτόμαστε ότι άλλες χώρες θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν άμεσα προς τις αξίες μας είναι κάπως υπερφιλόδοξο. Πρέπει πράγματι να ανοίξουμε ένα διάλογο, μια ανταλλαγή πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική με ιδιαίτερη εστίαση στα θέματα των δικαιωμάτων και πράγματι οι διεθνείς εμπορική συμφωνίες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Εμείς θα επιχειρήσουμε λοιπόν να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τις εισηγήτριες για να βρούμε ένα κοινό έδαφος. Διότι όπως σήμερα υποβάλλεται το σχέδιο, θα είναι πολύ δύσκολο για το ΕΛΚ να το υποστηρίξει. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, thank you very much and I turn Ευχαριστώ και τώρα... Ε, ε, επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ. Από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πάντα υπό το πρίσμα της διαφοράς ανδρών και γυναικών. Αυτό βεβαίως ε, είπε ο συνάδελφος, αλλά πρέπει να πω ότι η εμπορική πολιτική ε, αυτή τη στιγμή πραγματικά ε, υποσκελίζει τη, την, τη διάσταση ανδρών γυναικών και πρέπει στο μέλλον το αλλάξουμε αυτό. Να σκεφτούμε πώς οι συμφωνίες αυτές επηρεάζουν την κατάσταση των γυναικών, όχι μόνο στις χώρες μας, αλλά και στις χώρες με τις οποίες συνάπτουμε τις συμφωνίες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η διάσταση και διαφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Ε, δεν είναι βεβαίω οι γυναίκε ένα μόνο μπλοκ. Ε, είναι καταναλώτριε, είναι γεωργοί, ε, έχουν κάποιο εισόδημα ή δεν έχουν, είναι νοικοκυρέ. Σε όλου αυτού του διαφορετικού ρόλου οι επιπτώσει ποικίλουν. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα στην έκθεση. Όπως και να έχουν τα πράγματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εργάζομαι και στην Επιτροπή Γεωργίας, στις εμπορικές συμφωνίες πουθενά δεν αναφέρονται στο θέμα ε, της βιώσιμης γεωργίας, ε, του ύδατος, των σπόρων, ε, της ε, καταπάτησης των πόρων της γης, δεν έχει ληφθεί υπόψη εκεί λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των πόρων σε πολλές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε οι εμπορικές συμφωνίες να μην οδηγήσουν σε διαδικασίες συγκέντρωσης ε, πλούτου και να μην όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκλεισμένοι από αυτούς τους πόρους. Και μια κακή εμπορική πολιτική ε, μπορεί να έχει αποτέλεσμα μεταναστευτική πίεση. Και αυτό συμβαίνει. Και λυπάμαι που δεν το λέμε και πιο ειλικρινά. Όταν ακολουθούμε μια λαθασμένη εμπορική πολιτική, το αποτέλεσμα στην άλλη πλευρά του κόσμου είναι ροές, μεταναστευτικές ροές. Και αυτό βεβαίως έχει επηρεάζει διαφορετικά και περισσότερο τις από τους άντρες. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην έννοια αυτή των εθελούσιων συμφωνιών. Διότι λέμε συχνά ότι οι εμπορικέ συμφωνίε ε, συνάπτονται ε, εθελοντικά ε, από τα κράτη-μέλη, με τη βούλησή τους δηλαδή. το θέμα είναι όμως Ποιο έχει λόγο σε μια χώρα όταν συνάπτεται μια εμπορική συμφωνία. Οι γυναίκε δεν βλέπω ποτέ στην τραπέζι διαπραγματεύσεων σε τέτοιου είδου συμφωνίε οι γυναίκες ε, συμμετέχουν τελικά στην, ε, στο σχεδιασμό μιας εμπορικής συμφωνίας και στη σύναψή της. Ε, όταν έχουμε μια διαφήμιση στην Γερμανία κάποιο νέο φάρμακο, ε, συχνά υπάρχει μια προεδοποίηση που μιλάει για τις παρενέργειες και όταν υπάρχουν παρενέργειες πηγαίνετε να δείτε το φαρμακοποιό σας. Εδώ προσπαθούμε τις εμπορικές συμφωνίες ε, να δούμε ποιες είναι οι παρενέργειές τους στις γυναίκες. Και αυτό επίγει. Δεν συμφωνώ καθόλου ότι ε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεπεράσει. Όχι. Είναι μια νέα προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε ό,τι την εμπορική ε, πολιτική μας. Είναι καλό που γίνονται αυτές οι κοινέ συνεδριάσεις με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, με την Επιτροπή Γυναικών, διότι αυτά τα θέματα, θέματα είναι οριζόντια. Αφορούν πολλές επιτροπές και πρέπει να οικειοποιηθούμε αυτά τα ζητήματα από κοινού. Θέλω να ευχαριστήσω για την συνεδρίαση αυτή την κοινή. Ευχαριστώ πολύ. η συγγήτρια από το ECR, από την Επιτροπή Γυναικών, δεν είναι εδώ, από το ALDE, από το EFDD, ENF, α, συγγνώμη, η συνάδελφος Τιτσιάνα Μπεγκίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δίνουμε στην ΙΝΤΑ και ε, για τη συνάδελφο Ντανιέλα Γιούτο ε, θα πρέπει να εργαστώ για την, ε, το βραβείο Σαχάροφ. Και συνεχίζω Ιταλικά. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ τις εισηγήτρες για την εξαιρετική τους δουλειά. Πράγματι η εμπορική πολιτική είναι το πιο ισχυρό μέσο που έχουμε στη θέση μας ώστε να επιβάλλουμε τον σεβασμό προ τα θεμελιώδη δικαιώματα για την ισότητα των φύλων. Αυτό πρέπει να είναι σαφέ για του νομοθέτε, πρέπει να είναι σαφέ και για του διαπραγματευτέ τέτοιων συμφωνιών και πρέπει να είναι σαφέ ότι όταν μιλούμε για αντίκτυπο των συμφωνιών αυτών επί ε, των θεμάτων ισότητα, πρέπει να έχουμε κατά νου μια αμυντική σκοπιά και μια επιθετική. Καταρχά, οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών δεν πρέπει να έχουν αρνητικέ συνέπειε άμεσα ή έμεσα στις γυναίκε και τα δικαιώματά τους. Πρέπει να υπηρεσπιζόμαστε του πολίτες μας. Όπως σωστά λένε οι συγκήτριες, η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή βασικών αγαθών όπως το νερό μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία τους αλλά και στην πρόσβαση και στην ομαλή τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι η αμυντική πτυχή της οποία θα θέλαμε θα προτείνουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Από την άλλη μεριά πρέπει και να είμαστε πιο ενεργητικοί, πιο επιθετικοί αν θέλετε. Να μην σκεφτόμαστε μόνο την άμυνα αλλά και την επίθεση για την προαγωγή μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Επομένως δηλαδή να εισαγάγουμε ρήτρε δεσμευτικές στις συμφωνίες αυτές, σαφή σχετικά με την επιβολή των μέτρων για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της άτυψης και να ζητούμε πιστοποιήσεις για τα διάφορα αγαθά που διέπουν οι συμφωνίες αυτές ως προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς οικονομίας όπως την κλωστοϊφαντουργία έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των γυναικών αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο το οποίο τις καθιστά πολύ πιο ευάλωτες σε εκμετάλλευση, σε παραβιάσεις, σε προκλήσεις, το οποίο ισχύει και για τον γεωργικό τομέα. Και όπως είχα πει και την περασμένη φορά που συζητήθηκε το θέμα, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να διοργανώσουμε ανταλλαγές πολιτιστικών απόψεων και κοινοπραξιών μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες στις χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Αυτή τη στιγμή μόνο ένα στα πέντε κεφάλαια αναφέρονται στα θέματα αυτά. Οι μελλοντικέ λοιπόν συμβάσει θα πρέπει να ενέχουν αυτά τα αμυντικά και επιθετικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε αμέσω γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Ε, thank Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και τώρα στρέφομαι στις σκιώδεις συγκητές της ΙΝΤΑ. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου που αντιπροσωπεύω από Σαΐφη που είναι ε, σκιώδης εισηγήτρια για το ΕΛΚ αλλά δεν μπορεί να είναι παρούσα. Ε, ευχαριστώ τις εισηγήτριες για το σχέδιο έκθεσης που διαβάστηκε από τη συνάδελφη και Υπάρχουν ε, μερικές προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Βλέπουμε το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες ως μέσο προώθησης της οικονομίας και για τις γυναίκες επαχειρηματίες στον εμπορικό τομέα. Αυτή είναι μια ιδέα που δεν περιλήφθη στην εισήγηση και είναι σημαντικό να τονιστεί η ιδέα αυτή. Υπάρχει ένα ε, σημαντικό δεδομένο 40% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήκουν σε γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να εξακολουθήσουμε να έχουμε υποστηρικτικά μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σύσταση για την διαπραγμάτευση του εξυγχρονισμού ε, του, του εμπορικού πυλώνα ε, για, στην συμφωνία με τη Χιλή ζήτησε να περιληφθεί η ευτονομία των γυναικών και η ισότητα των φύλων και ελπίζουμε η συζήτηση θα ακολουθήσει αυτόν τον προσανατολισμό και θα συνοδευτεί με άλλα μέτρα. Σχετικά με το σχέδιο εισήγησης είναι σαφές ότι το ΕΛΚ θα υποβάλει τροπολογίες για οι ορισμένες ιδέες να συμπληρώσει την εισήγηση. Θα θέλαμε να τονίσουμε την έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών για τα θέματα του εμπορίου και των επιπτώσεων επί της ισότητας των βήλων. Και λυπούμεθα ότι ε, το, το θέμα της ισότητας των βήλων δεν περιλαμβάνεται ε, στην μελέτη αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να περιλάβει ε, στις ε, μελλοντική στρατηγική ε, το θέμα της ισότητας των φύλων και να περιληφθεί επίσης τον προβληματισμό για την παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε να ενισχύσουμε το σίγμα γάμα πι συν ένα και υπάρχουν ήδη δύο θέματα σχετικά, σχετικά με την εξάλληψη όλων των μορφών ε, διακρίσεων κατά των ε, γυναικών και για την ίση αμοιβή. Το Κοινοβούλιο πάντοτε υπερασπίστηκε στα ψηφίσματα το θέμα ε, του αποκλεισμού των γυναικών είναι από, τα, από τις γραμμές. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με το θέμα σε διεθνές επίπεδο και μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ για να υπάρχει μια δυναμική ισχυρή για το θέμα αυτό. Τέλος, θα θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα της εισαγωγής των διατάξεων για τη νησότητα των φύλων, την συνεκτίμηση του θέματος, ειδικά κεφάλαια στις συμφωνίες που θα ασχολούνται με μέτρα λεπτομερή και δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως είχαμε τα σχόλιά σας και βεβαίως ε, μοιράζουμε τα όσα είπε η Μπάρμπαρα Ματέρα διαμέσου της αντιπροσώπου της. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες. Αυτή ήταν ε, η παρέμβαση εκ μέρους της ε, Ισάια Σαΐφη και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σοσιαλιστές εκ μέρους της. Είμαι, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες ε, για το σχέδιο εισήγησης. Θα πρέπει να δώσουμε όθηση, να έχουμε πλήρη πρόταση για το πώς να προωθήσουμε την ισότητα στο εμπόριο ε, και το, θα πρέπει ε, το είδαμε ότι η Κομισιόν, ο ΠΟΕ και μερικά κράτη-μέλη ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Επίσης, η ITC ε, κάλυψε 20 ε, αναπτυσσόμενες χώρες και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει επίπτωση πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο εμπόριο και προσπαθούν να εξαλείψουν τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην συμμετοχή ε, στο εμπόριο έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις, στην πληροφορία, στη χρηματοδότηση. Η ομάδα μου, σοσιαλιστές και δημοκράτες, υποστηρίζουμε πολλούς από τους στόχους του σχεδίου. Υπάρχει ανάγκη να περιλάβουμε την διάσταση του φύλου στην πολιτική, να υπάρχουν ε, κεφάλαια και να έχουμε μέτρα ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης να θεωρήσουμε και κυρώσεις που υπάρχουν ε, και στο, στην συμφωνία TTIP. Επίσης θα υποβάλω τροπολογίες για να ενισχύσουμε τους κοινού μας στόχους. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ευαίσθητη στην ισότητα των φύλων. Αυτό που άρχισε ο ΠΟΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, δραστήριες πολιτικές για την, για εξάλληψη των διακρίσεων και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αντιπροσώπευση των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί στους θεσμούς που διαπραγματεύονται. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε δεδομένα, στοιχεία χωριστά ε, για τα φύλλα και ε, για κάθε στρώμα της κοινωνίας. Βεβαίως όλες οι γυναίκες ε, δεν ξεκινούν από την ίδια δομή την κοινοοικονομική. Το κεφάλαιο για τις γυναίκες και το εμπόριο που θα πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης για την ΤΙΣΕ και ε, την τελευταία εβδομάδα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού είδαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο για τις εμπορικές ε, συμφωνίες και να διευκολύνουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ενίσχυση των εικονοτήτων των μέσων, ε, την πρόσβαση στις δημόσιους διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις για το σκοπό αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά εργαλεία και επίσης την Συμφωνία Διευκόλυνσης του ΠΟΕ. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την διάσταση του φύλου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα σκιώδης ηγητής από το ECR, από τους φιλελεύθερους, από τους πράσινους. Όχι, θέλω να κάνω κάποια προσωπικά σχόλια, αλλά όχι ο σκιώδης. Ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Πρώτα ε, θα ζητήσω να πάρουν το λόγο οι Σκιώδης και μετά και οι συνάδελφοι, οι ευρωβουλευτές. Το EFTD μίλησε ήδη, η ΕΝΕΦ δεν βλέπω κάποιο θέλει το λόγο. Τώρα απευθύνομαι στους ευρωβουλευτές γενικότερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα να σας πω δύο λόγια στο όνομα της Μαρία Ρώμα που δεν είναι εδώ σήμερα. Εκπροσωπώ τρία άτομα ουσιαστικά εδώ. Η Μαρία Αρένα ε, θεωρεί ότι σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες αυτές οι πολιτικές δεν παρουσιάζουν κανένα πλεονέκτημα. Αυτές οι συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών έχουν μόνο μειονεκτήματα για τις γυναίκες. Τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι σεβαστά, οι γυναίκες ε, είναι προϊόν εκμετάλλευση στη γεωργία, στην κλωσταϊφαντουργία, υπάρχει το θέμα της αρπαγής της γης, ε, η κυρία Αρενά θα ήθελε να ξέρει αν μπορούμε να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών έχουν επιπτώσεις στις γυναίκες παγκοσμίω. Ε, και αυτές οι επιπτώσεις είναι συνήθως αρνητικές. Στον τομέα της βιομηχανίας μπορεί να υπάρχουν κάποια ωφέλη, αλλά αυτά τα ωφέλη αφορούν τους άντρες στον τομέα των μεταφορών παραδείγματο χάρη. Η Μαρία Αρενά αναφέρεται ιδιαίτερα στον κλωστιφαντουργικό ε, κλάδο ποιες είναι επιπτώσεις δηλαδή της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων προς χώρες με χαμηλότερο εργατικό κόστος, σε ποιο βαθμό οι γυναίκες πλήττονται από αυτό το φαινόμενο. Τώρα προσωπικά θα ήθελα και εγώ να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη διαπραγμάτευση ό,τι αφορά το σχέδιο ψηφίσματος για τη συμφωνία με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Η εντολή διαπραγμάτευσης ε, θα καθοριστεί από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Καλό θα ήταν να εκφραστείτε εκεί ε, και, στο θέμα, και γύρω από το θέμα τη ισότητα των ανδρών και γυναικών. Είμαστε σε συντονισμό με τον κύριο Γκασπαρίνη ε, με τον κύριο Γκασπάρη για να γίνει ρητή αναφορά ε, τη σχέση ανδρών και γυναικών. Ε, ο κ. Γκασπάρη συμφωνεί, όμω στην πλευρά του ΕΛΚ και του ECR ε, δεν υπάρχει και ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ούτε πλευρά του Φιλελευθέρων. Υπάρχει όμω μια ολόκληρη νέα γενιά η οποία στηρίζει αυτήν την διάσταση και θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσεί να πείσετε του συναδέλφου σα ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα τέτοιο κεφάλαιο που θα αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και βεβαίω θα χρειαστεί πλειοψηφία για να συμβεί κάτι τέτοιο. πρέπει να ορίσουμε ποιε θα είναι οι δυνατότητε που θα έχουν οι γυναίκε στα πλαίσια αυτών των, των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών. Έω τώρα λίγα δεδομένα έχουμε στη διάθεσή μα, εξού και η πρότασή μα. Ο στόχο μα είναι λοιπόν να συλλέξουμε δεδομένα που θα μα ε, επιτρέπουν να προσμετρήσουμε τι επιπτώσει για τι γυναίκε όταν υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε και πώ μπορούν να αποφεληθούν πραγματικά από αυτέ. Ε, καλό θα είναι λοιπόν να μπορέσετε να πείστε του συναδέλφου σα έτσι ώστε ένα τέτοιο κεφάλαιο να συμπεριληφθεί στι συμφωνίε ευθύνων συναλλαγών με την Αυστραλία και την Νέα Λοιπόν, δύο πράγματα πρέπει να κάνω. Πρώτα πρέπει να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο ο οποίο θέλει το λόγο. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα πρέπει να απαντήσω όμως τώρα ε, στην έκκληση. Και θέλω να υπενθυμίσω ε, βεβαίως ε, στους συναδέλφους και εγώ διάβαζα αυτά που μου είπε η Τοκία, η Τοκιά. Με αυτήν θα συζητήσετε. Εάν θέλετε τη δική μου άποψη, η άποψή μου είναι διαφορετική από αυτά που διάβασα. Έτσι. Εγώ εδώ εκπροσωπούσα τη συνάδελφο, την κυρία Σαϊφή. άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που άκουσε, που είπε ο συνάδελφος πάλι στο όνομα του συνάδελφου, συνάδελφου Ματέρα αυτό είναι πιο κοντά και στις δικές μου απόψεις, ένα από τα ζητήματα στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι το εξής. Το εμπόριο είναι όντως ένα όχημα ε, για πολλές από τις πολύ σημαντικές αξίες της Ένωσης. Είναι ένα όχημα και οι εμπορικές συμφωνίες προωθούν αυτές τις αξίες. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε, εν ότι οι εμπορικέ συμφωνίε αφορούν το εμπόριο. Εάν δηλαδή φορτώσουμε πολλού άλλου στόχου στι εμπορικέ συμφωνίε, αυτό θα καταστήσει πολύ δύσκολη τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών στο μέλλον. Βεβαίω πρέπει να προσπίσουμε τι βασικές αξίε της Ένωσης, αλλά το ΕΛΚ πάντα ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για το τι πρέπει να συμβεί και τι μπορεί κυρίως να συμβεί και πραγματικά με τιμά το γεγονός ότι ε, η συγγήτρια αναφέρθηκε στην έκθεση ε, για τις ε, διενέξεις ήταν ένας τρόπος ε, να προσεγγίσουμε διαφορετικά τα προβλήματα του κόσμου και να πω ότι συχνά στην Επιτροπή αυτή, στην έκθεση αυτή, είπαμε ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα που προκύπτουν ε, στις ζώνες σύραξης ε, ε, της καταχρήσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τους εμφύλιους πολέμου, να τα λύσουμε αυτά με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, διότι δεν είναι προβλήματα εσωτερικά της Ένωσης. Συμβαίνουν εκεί αυτά. Ένας κανονισμός είναι απλά ένα εργαλείο που συνδυαζόμενο με άλλα εργαλεία, η πολιτική ανάπτυξη, πρέπει σίγουρα να, την μεταρρυθμίσουμε σημαντικά η ενίσχυση για το εμπόριο ε, έτσι ώστε αυτές οι χώρες να γίνουν πραγματικά κράτη δικαίου διότι κάποια κράτη από αυτά δεν λειτουργούν ε, ε, δεν μπορούμε να επιλύσουμε όμως τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιληθούν εφόσον εμείς τους ε, δώσουμε κάποια εργαλεία που θα τους βοηθήσουν και κάποιες βεβαίως δεσμευτικές ε, ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη η παρουσία μας εκεί. Αυτά θα δώσω τώρα το λόγο στη Συμπρόεδρο. But I would like to Βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε και την κυρία Μπιόρκ για τα τελικά της σχόλια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο Πρόεδρους πάντα είναι ωραίο να επισκέπτεται κανείς και άλλες ε, επιτροπές, να ακούει και άλλες προσεγγίσεις και οπτικές. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο θα μας διαφωλύνει ε, να υπερασπιστούμε των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει να έχουμε αιτήματα, γιατί είναι οικονομικό ζήτημα στο οποίο μπορούμε να έχουμε επιρροή, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που θα έχουμε διάθεσή μας γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε κάποιες διαφορές προσέγγισης, αλλά πολλοί από τους συναδέλφους μου εδώ και στην Ίντα και στην Επιτροπή Γυναικών έχουν τοποθετήσει αυτά στο σωστό τους πλαίσιο, στην ανάγκη για δεσμευτικούς κανόνες και διατάξεις, ίσως και στην ανάγκη κυρώσεων στα πλαίσια των συμφωνίων αυτών, Δηλαδή τι κάνουμε όταν οι εταίροι μας δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες από τον οποίο έχουμε συμφωνήσει στα θέματα των δημοσίων υπηρεσιών που είναι πάρα πολύ σημαντικά υπό την έννοια της ισότητας των φύλων γιατί έχουμε διάφορες ομάδες γυναικών και διάφορες ιδιότητες τους ως καταναλωτές, ως πολίτες κτλ. Και πρέπει να ενσωματώσουμε όλες τις πτυχές αυτές. Όμως, πρώτα απ' όλα έχουμε μια επίκαιρη, έγκαιρη γνωμοδότηση σε στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή ε, υποβάλλει πρόταση σχετικά που θα διέπει δηλαδή τις διεθνείς συμφωνίες και πρέπει αυτό να το κάνουμε και να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Βλέπω και ακούω τα σχόλια σχετικά με το δεσμευτικό κεφάλαιο, κεφάλαιο. Άκουσα και τα σχόλια της συναδέλφου για τα στοιχεία επιθετικής πολιτικής που πρέπει να έχουμε, τακτικής, αλλά και αμυντικής. Επομένως, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον όλες σας τις προτάσεις τροπολογιών. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η πρόεδρος θα μας πει ποια είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών, αλλά περιμένω να τα δω όλα αυτά γραπτός με μεγάλο ενδιαφέρον για να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή. Και ευχαριστώ και για τη συνεισφορά της στην συνεισηγήτρια κυρία Φορέντσα που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Η προθεσμία 16 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Δεν έχουμε. Έχουμε λίγες μέρες. Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση και σας ευχαριστώ κύριε Βίνκλερ η επόμενη ε, συνεδρίαση 22 Νοεμβρίου για την εξέταση των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Έληξε η συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και οι διερμηνείς ευχαριστούν την πρόεδρο και ευχαριστώ την γραμματεία για την προετοιμασία της συνεδριάσεώς μας.